Κυρίε Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσω στην μητρική μου γλώσσα, τα τσεχικά. Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε τη δήλωση της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Θα σας παρακαλούσα. Επίτροπε, έχετε το λόγο. The new coming, uh, new... Πρόεδρε, ε, η κατάσταση